ευρύτατη ε, συνένεση στο Κοινοβούλιο ε, και ότι θα περάσει το κείμενο αυτό μεγάλη υποστήριξη στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ολοκλώθηκε το σημείο αυτό της μισή διατάξεως. Θα ψηφιστεί σήμερα στις 12.00. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Προφορικές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις ομάδες των εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής ε, και την ισορροπημένη εκπροσώπηση καθώς επίσης και τη διαφάνεια. Υπάρχουν ε, προφορικές ερωτήσεις. Ο κύριος Ντε έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Επιτροπή πέρσι αναθεώρησε τους ε, κανόνες που διέπουν τις ομάδες εμπειρογνωμόνων Έκανα πολύ καλέ ανεπίσημε συζητήσει με του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, είναι περίεργο το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ποτέ επίσημα δεν συμμετείχε, γιατί η διαφάνεια απασχολεί τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και την Επιτροπή. Μπορούμε να με διασφαλίσει ότι ο Επιτροπό ότι στο μέλλον θα γίνεται για τέτοια θέματα επίσημο διάλογο προτού λαμβάνονται οριστικέ αποφάσει τις προηγούμενες εβδομάδες ε, ήρθα σε επαφή με διάφορες ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και δυστυχώς ε, ανησυχούν ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ομάδες εμπειρογνωμόνων και την ισορροπημένη εκπροσώπησή τους. Και μιλάμε κυρίως... Να σας πω ότι η δική μου εμπειρία ήταν ότι οι γενικές διευθύνσεις είναι μικρά βασίλεια. Αλλά αν υπάρχει πολιτική θέληση θα πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχει ένα κοινό, μια κοινή ιστοσελίδα για τους εμπειρογνώμονες και για να υπάρχει και μια ενιαία διαδικασία καταχώρησης. Θα αναλάβει δράσεις εδώ ο Επίτροπος, όλες ε, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα συνδικάτα, οι ενώσεις καταναλωτών, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει να συμμετέχουν με ένα μικρό γραφείο στις Βρυξέλλες. Αυτό σε αντίθεση με τις μεγάλες εταιρείε που έχουν ειδικά τμήματα. Αυτό τι σημαίνει ότι τα συμφέροντα των καταναλωτών, των πολιτών, των ανθρώπων που δεν είναι ε, στις Βρυξέλλες ε, ε, δεν εκπροσωπούνται παρκώς. Και αυτό συνεπάγεται και ένα κόστος. Θα πρέπει να διευκρινίζεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ε, αποζημιώνονται τα έξοδα αυτά διαμονής και ταξιδίων. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει συχνά δεν γνωρίζουν ότι επιστρέφονται τα έξοδα αυτά και δεν ε, το υποδεικνύουν αυτό πάντα οι υπάλληλοι της ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Για ένα μικρό αυτοαπασχολούμενο δεν είναι δυνατόν να αφήσει τη δουλειά του και να ταξιδέψει και να μείνει στις Βρυξέλλες. Χρειάζονται την αποζημίωση των εξόδων. Η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ θεωρεί ότι οι εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν προσωπικά δεν έχουν σχέσεις με οργανώσεις που ε, είναι άμεσα συνδεμένες με τα συμφέροντα της ομάδας εμπειρογνωμονών. Καλό λοιπόν να συνδεθούν οι γενικέ διευθύνσει μεταξύ του. Να μας πει ο Επιτροπός επίσης πώς είναι ο δυνατόν να αναφέρεται στην ισοσελίδα της Επιτροπής η Greenpeace ονομαστικά σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της πλατφόρμας τεχνολογίας ενώ κατέχω αλληλογραφία μεταξύ της Greenpeace και της ε, Επιτροπής ενώ φαίνεται ότι από την οποία προκύπτει ότι δεν επιτρέπει και η συμμετοχή στην Greenpeace. Ευχαριστώ για δύο λεπτά. Το λόγο έχει ο κ. Κάσουμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Καλώ ήρθατε στον κόσμο τη πολιτική, όπου κανεί δεν ενδιαφέρεται σε αυτά που πετυχαίνει σωστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο ενδιαφερόμαστε που κάνετε λάθο. Είναι πολύ καλή η πρωτοβουλία, αλλά το Κοινοβούλιο, όπω είπε ο κ. Ντεγιόνγκ, έχει κάποιε ανησυχίε. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι ομάδε εμπειρογνωμόνων είναι ανοιχτέ και μπορούν να συμμετάσχουν και ευρύτερε ομάδε και να έχουν το έξω πληροφορίε ε, όσον αφορά την πρόσβαση στι ομάδε εμπειρογνωμόνων. Θέλουμε να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη στις ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων. Για να γίνει αυτό χρειάζεται απόλυτη διαφάνεια και όπως υπόθηκε δεν πρέπει να επικρατήσουν μεγάλες επιχειρήσεις. Αλλιώς θα υπάρχει κατηγορία ότι υπάρχουν συμφέροντα και αυτό υπονομεύει το έργο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το έργο των ομάδων εμπειρογνωμών. Και το λέω σαν εισηγητή όσον αφορά τον αρχικό κανονισμό για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που εφαρμόσαμε στο Κοινοβούλιο του 2001. Όπω τα ξέρετε, Επίτροπε, η όλη αρχή τη ανοιχτή προσέγγιση και λήψη αποφάσεων κοντά στου πολίτε όσο είναι δυνατόν αυτόν απορρέει τη συνθήκη του Άμστερνταμ και αυτό το εφαρμόσαμε με τον κανονισμό 1049-2001. Αυτό είναι κάτι που αναθεωρείται όμως τώρα και είναι μια καλή ευκαιρία πιστεύω για το πρόγραμμα πλαίσιο για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων να εισαχθεί στην αναδιατύπωση του κανονισμού, στην πρώτη σχετική που δεν δέχεται το Κοινοβούλιο, την πρώτη του 2008. Όπως θα παρατηρείτε η κυρία Μακοβέ είναι στην αίθουσα, έχει μακρά ιστορία ζητώντας μεγαλύτερο άνοιγμα και διαφάνεια και οι περισσότερες πολιτικές ομάδες δίνουν μεγάλη σημασία στο θέμα. Θα ήθελα να ξέρω γιατί το Κοινοβούλιο δεν έξαβα στην άποψή του. Θα έχετε ε, μια ιστοσελίδα για καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για το πώς οι εκπρόσωποι των πολιτών και, και οι οργανώσεις των πολιτών μπορούν να συμμετάσχουν με καλύτερο τρόπο. Αλλά όπω είπα στην αρχή, καλώ ήρθατε στον κόσμο τη πολιτική όπου όλοι έχουν μανία με τι ελλείψει παρά με τα επιτεύγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κάσμαν. Για δυόμιση λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Καμφά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, καλημέρα Επίτροπε συμμετέχω συντάξει σε αυτήν την ερώτηση, διότι θεωρώ ότι είναι υψή τη σημασία τόσο για την Κομισιόν αλλά όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολότη να είναι καταστεί διαφανή στο θέματα των ε, lobbying και τη άσκηση επιρροή. Ξέρετε ότι στι Βρυξέλλε υπάρχουν περισσότεροι λομπίστε από όλη την Ουάσιγκτον. Και ένα τρόπο για να ασκήσουν την επιρροή του ε, παρά την Επιτροπή είναι αυτέ οι ομάδε προγραμμών. Εγώ συμμετέχω στην Επιτροπή Νομισματικών και Οικονομικών Θεμάτων. Έχετε μια ομάδα ε, εμπειρογνωμών στα θέματα ε, τραπεζικά. Το 80% αυτών των συμμετεχόντων είναι τραπεζίτες και τραπεζίτες των επενδυτικών μεγάλων ομίλων, Goldman Sachs ε, κλπ. Δεν υπάρχει μια κυβερνητική εκπροσώπηση, δεν υπάρχουν συνδικάτα σε αυτή την ομάδα των πυρογνωμόνων. Η ιδέα του να ε, συμβουλεύεται η Επιτροπή μόνο ε, τέτοιου είδους εμπειρογνώμονες θεωρώ ότι είναι κάτι το σουρεαλιστικό μετά από την οικονομική κρίση που γνωρίσαμε. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα σημεία σε αυτή την προφορική ερώτηση που σας ε, θέτουμε. Θα αλλάξετε τη σύνθεση ε, αυτών των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Θα φροντίσετε ούτω ώστε τα πρακτικά να δημοσιοποιούνται υπό σύγκρουση συμφερόντων να αποφεύγεται. Φυσικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό είναι ζήτημα ε, διακομματικό. Υπάρχουν ε, ε, φιλελεύθεροι, πράσινοι, δεξιοί, οι σοσιαλιστές που ενδιαφέρονται γιατί λοιπόν δεν φροντίσατε να συμβουλευτείτε και το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Καμφέν για δυόμιση λεπτά. Το λόγο έχει η κυρία Λεπάζου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, συμφωνώ 100% με τους προλήσαντες συναδέλφους και ιδιαίτερα με τον κύριο Ντεγιόγκ και τον κύριο Καμφέ δεν μπορώ παρά να εκφράσω την λύπη μου που το Κοινοβούλιο δεν συμμετείχε στις διαδικασίες προκειμένου να ληφθεί μια σωστή απόφαση. Αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί σε τακτά διαστήματα, ειδικά στο πλαίσιο της Επιτροπής Υγείας και Περιβάλλοντος, όπου έχω και εγώ μια εμπειρία παρόμοια με αυτή που εξέφρασε ο συνάδελφος Πασκάλ Κομφέ. Θα ήθελα και επίτροπε να επιμείνω επί δύο σημείων. Το, στην ισορροπία των ομάδων είναι ζήτημα πολύ σημαντικό έχουμε μια σύνθεση ιδιαίτερα ανισομερή, πάρα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις, ελάχιστες μικρές, βιομηχανικός κλάδος και όχι η κοινωνία των πολιτών. Αυτό λοιπόν το βάρος των ομάδων έχει ε, σημαντική βαρύτητα στις αποφάσεις που λαμβάνει η Κομισιόν διότι στηρίζει τις αποφάσεις της, της ε, γνώμης των εμπειρογνωμόνων. Ως εκ τούτου, όπως καταλαβαίνετε, η επανεξισορρόπηση υπέρ μιας ε, μεγαλύτερης εκπροσώπησης της κοινωνίας των πολιτών είναι κάτι το απαραίτητο και στους νέους τους κανόνες δεν βλέπουν προτάσεις ούτε υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ούτε υπέρ της κοινωνίας των πολιτών. Το δεύτερο ερώτημα είναι αυτό της ε, επιλογής των εξωτερικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων. Είναι απολύτως απαραίτητο να γνωρίζετε και να γνωρίζουμε ποιος μιλάει και εξ ονόματος ποιου. Όταν ένα εμπειρογνώμων ε, ε, εμφανίζεται ως ε, ανεξάρτητος ενώ είναι φορέας lobbying δεν μπορεί να γίνεται δεκτός τη συμμετοχή σε αυτές τις ομάδες εμπειρογνωμόνων. Είναι απαραίτητο λοιπόν ο έλεγχος και των, των δηλώσεων συμφερόντων να γίνεται αποδεσματικά. Χρειάζεται να γνωρίζουμε λοιπόν κατά πόσον παρεμβαίνει ως ε, καθηγητής θα λέγαμε ενώ στην ουσία εκπροσωπεί μια βιομηχανία τα πράγματα δεν είναι σαφή θεωρώ λοιπόν ότι η σύγκρουση συμφερόντων είναι πολύ σημαντικό ζήτημα έχουμε μια νέα απόδειξη με ένα σοβαρό πρόβλημα στην υπηρεσία φαρμάκων και θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε ως εκ τούτου λοιπόν κύριε Επίτροπε σας ζητητεύω φροντίστε να ε, αποκτήσουμε εκ νέου εμπιστοσύνη στους εμπειρογνωμόνες που χρησιμεύουν ως ε, βάση στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Ευχαριστώ κύριε Αλεπάζου. Το λόγο έχει ο Επίτροπος κύριος Κάλλας. Σας ευχαριστώ πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Φυσικά δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζετε το ιστορικό υπόβαθρο του θέματος αυτού, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα που αντικαθιστώ τον συνάδελφο Σεφκοβιτς και που απαντώ στο ερώτημα αυτό για τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν δικός μου ο τομέας αυτός. Ήμουν αρμόδιος σε τέτοια θέματα και φυσικά χαίρομαι που μπορώ να σας πω τι άλλαξε πραγματικά. Και οι ομάδες εμπεριγνωμόνων πώς τροποποιήθηκαν. Και δυστυχώς έχω τρία λεπτά μόνο να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Όπως αναφέρατε υπάρχει ένα νέο πλαίσιο το οποίο εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2010 για τους εμπειρογνώμονες και ε, προβλέπει ότι όταν ορίζεται η σύνθεση των ομάδων αυτών τα τμήματα της Επιτροπής θα προσπαθούν να υπάρχει ίση εκπροσώπηση σε ό,τι αφορά και τις τομείς ε, εμπειρογνωμοσύνης, λαμβάνοντας υπόψη και τις εργασίες που θα πρέπει να γίνουν και τις εμπειρογνωμοσύνης που χρειάζεται το νέο πλαίσιο προβλέπει σαφείς και οριζόντιους κανόνες για να αποφευθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, οι αρμόδιες ε, υπηρεσίες της Επιτροπής θα ενημερώνουν τους εμπειρογνώμονες ότι αποδεχόμενοι να συμμετάσχουν στην ομάδα δεσμεύονται να βρουν ανεξάρτητα και υπέρ του κοινού συμφέροντας. Αυτοί οι κανόνες ισχύουν για όλες τις ομάδες εμπρευνομόδων και αποτελούν τη μία και μοναδική πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό. Τον Οκτώβριο του 2005 και αυτό μετά από καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον βουλευτών, ο Γιάννης Μπόντε ξεκίνησε ε, από την Επιτροπή ένα δημόσιο μητρό, το οποίο μας έδωσε με πληροφορίες για πολλά θέματα σε ό,τι αφορά τη σύνθεση και τα καθήκοντα των ομάδων από το 2007 και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σταδιακά δημοσίευε τη σύνθεση των ομάδων αυτών. Στο πλαίσιο του 2005 η αποκάλυψη μάλλον ε, της σύνθεση των ομάδων ολοκληρώθηκε το 2009. Άρα ουσιαστικά διατύφονται τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων στις ομάδες. Αυτό ήταν έντονη έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2005 και πραγματοποιήθηκε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια ε, μια νέα έκδοση του Μητρώου το 2010, βελτιώνοντας τη διαφάνεια, παρέχοντας πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Για παράδειγμα, πιο πολλές πληροφορίες για τις οντότητες που συμμετέχουν και το καθεξής. Επίσης, μεγαλύτερη διαφάνεια για τις δραστηριότητες κάθε ομάδας, επιτρέποντας τις υπηρεσίες της Επιτροπής να δημοσιεύουν τέτοια στοιχεία ή να παρέχουν και ένα σύνδοσμο σε διάφορες ιστοσελίδες όπου μπορεί κανείς να βρει πιο πολλά στοιχεία. Δεδομένων των τεράστιου όγκου των πληροφοριών που έπρεπε να διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεχίζονται ακόμη οι εργασίες ε, για το Μητρό, άρα κάποια από τα δεδομένα θα πρέπει να επιβεβαιωθούν και η μετάβαση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες. Επιπλέον, επειδή επί 5,5 χρόνια πραγματικά συζητούσα τα θέματα αυτά με διάφορες ε, οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών και βουλευτές, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει απόφαση ότι είναι πολιτική ευθύνη της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρχει ίση εκπροσώπηση της ομάδας αυτός. Να μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε και αυτό το Μητρό Διαφάνειας ε, το 2005, το οποίο τότε αναφερόταν ως Μητρό Λόμπι και τώρα γίνονται προσπάθειες να γίνει, υπάρχει και ένα κοινό μητρό με το Κοινοβούλιο. Άρα τα πράγματα βελτιώνονται, δεν πάνε και άσχημα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Περνάμε τώρα στους ομιλητές εξονόμενων των πολιτικών ομάδων. Το λόγο έχει η κυρία Μακοβέη, εξονόμενος του Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπε για την απάντησή σας και χαίρομαι που παίρνω το λόγο μετά από εσά. Θα ήθελα να πω ότι καλύτερα να κοιτάμε το παρόν και το μέλλον παρά το παρελθόν και καλύτερα να δούμε μεγαλύτερα βήματα προς τη διαφάνεια. Συμφωνώ με τους συναδέλφους όσον αφορά το θέμα αυτό και υπενθυμίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει δράση τόσο ώστε να υπάρχει ισόρροπη εξορρόπηση των διαφόρων ομάδων συμφερόντων στη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Όπως αναφέρατε έχουμε ένα θεωρημένο πλαίσιο αλλά απομένουν πολλά προβλήματα κατά την άποψή μας που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη του κόσμου. Και θα αναφερθώ σε κάποιες ελλείψει οι διαδικασίε για τον τοπισμό και εξάλληψη σύγκρουσεων συμφερόντων λείπουν. Χρειάζονται διαδικασίε για να εντοπίζονται και να εξαλείφονται αυτέ. Δεν αρκεί να στέλνουμε επιστολή στου εμπειρογνώμονε και να μα πούν αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ή όχι. Ρήτρε όσον αφορά την επαγγελματική μυστικότητα ε, θα πρέπει να επεκταθεί από μέλη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέλη τη ομάδα ε, εμπειρογνωμών. Αντί κινούμεθα δηλαδή προ διαφάνεια, πάμε προ μεγαλύτερη μυστικότητα. Η έλλειψη διαφάνεια επιτροπη στα μελη τη ομαδα εμπειρογνωμων όσον μυστικοτητα η διαφανεια παραμενει οσον αφορα την ε, αποκάλυψη των εγγράφων που χρησιμοποιούν οι ομάδε εμπειρογνωμόνων. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει επίση και η κοινωνία των πολιτών και οργανώσει των πολιτών δεν εκπροσωπούνται σωστά. Ε, χρειάζονται μετά διαφυλάξει κατά τη επικράτηση τη βιομηχανία. Μπορεί τελικά οι μεγάλε επιχειρήσει να επηρεάζουν και να δεσμεύουν τι ομάδε εμπειρογνωμόνων. Θέλουμε περισσότερε πληροφορίε για τι υφιστάμενε αυτέ ομάδε εργασίε να θεθούν εγκαίρω στι σελίδε, οι πληροφορίε και τα μέλη των ομάδων και οι αιτήσει για τη συμμετοχή θα πρέπει να είναι διαφανείς και να αποκαλύπτονται. Επιμένω. Και όσον αφορά και τους πώ που πηγαίνουν σε δικαιούχος χρειάζεται διαφάνεια. Η διαφάνεια εξασφαλίζει ορθή διακυβέρνηση και εμπιστοσύνη εναντί των θεσμικών οργάνων. Αν θέλουμε ο λαός να έχει εμπιστοσύνη, αυτή είναι η μόνη λύση. Μεγαλύτερη, πλήρη διαφάνεια χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μακοβέη. Εξ των σοσιαλιστών για 1,5 λεπτό το λόγο έχει η κυρία Γκουρμάη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι, Επιτροπή. Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, ε, ανησυχίες για την ευρωπαϊκή λήψη αποφάσεων. Καταρχάς, ότι δεν είναι διαφανής η διαδικασία αυτή. Η διαφάνεια και η απλούστευση θα πρέπει να είναι οι δύο βασικές γραμμές για τη λήψη αποφάσεων σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε εδώ για να καταστήσουμε τη λήψη αποφάσεων πιο δύσκολη. Και δεν θα πρέπει να είναι ε, πάρα πολύ δύσκολη η πρόσβαση στις σχετικές ιστοσελίδες. Θα πρέπει να είναι φιλικές προς το χρήστη. Επίσης, ο ρόλος των λόμπι δεν είναι σαφής. Ο ρόλος των μεγάλων επιχειρήσεων είναι δυσανάλογα μεγάλος. Ξέρω ότι μπορεί να είναι χρήσιμο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί οι ομάδες πίεσης ε, είναι πάντα σημαντικές, αλλά πιστεύω ότι η διαφάνεια και πάλι είναι εκ των νουκ άνευ και ελπίζω να είμαστε πάρα πολύ ε, αποτελεσματικοί στο μέλλον σε ό,τι αφορά τις λίστες αυτές. Θα πρέπει να κοιτάμε τις ομάδες εμπειρογνωμόνων για αυτό που είναι, μια ομάδα που μπορεί να προσπίσει κάποια συμφέροντα. Αν δεν είναι αμερόληπτη συμμετοχή στις ομάδες αυτές, θα έχουμε άλλη ε, άλλο ένα πρόβλημα. Ωστόσο, αυτές οι ομάδες είναι, σωστά, είναι συνήθως επιτυχείς. Θα ήθελα λοιπόν να επαναλάβω τα, αυτά που ζήτησαν οι συνάδελφοι, να έχουμε ισορροπημένη εκπροσώπηση και αυτό είναι δεσμευτικό ή όχι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Γκουρμάη. Εξόρμαρο των σώμα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Γιόμπρο. Ο κύριος Γιόμπρο, συγγνώμη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι προφανές πως ε, σε κάθε κρατική κοινωνία η διαφάνεια θα πρέπει να είναι δεδομένη. Πρόκειται για μια προϋπόθεση για την ε, λήψη καλών αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψη πως ε, οι κοινωνίες ε, και οι οργανώσεις ενδιαφέρονται άμεσα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι οποιοσδήποτε ομάδες ή όργανα εμπειρογνωμών της Επιτροπής θα πρέπει να πετυχαίνουν την ισόρροπη εκπροσώπηση αλλά και την απόλυτη κατ' δυνατόν διαφάνεια. Είναι λοιπόν γεγονός ότι οι ομάδες των εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να λειτουργούν με βάση τους κανόνες της διαφάνειας προκειμένου να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων και δράσεις ε, που αποβαίνουν σε όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων. Ευχαριστώ πολύ για ένα λεπτό το λόγο ο κύριος Μπάτιν. Πέρσι τον Οκτώβριο το Κοινοβούλιο υπέβαλε έξι οδηγίες σχετικά με το θέμα. Στις 7 Φεβρουαρίου υπέβαλα μια προφορική ερώτηση στην Επιτροπή ε, ρωτώντας για ένα θέμα της πράξης για τις επιχειρήσεις του 76. Πρόκειται ε, για ένα παράδειγμα για μία επιχείρηση, δηλαδή την Τράπεζα της Αγγλίας. Αυτή η εξαίρεση, η παρέκκληση σχετικά ε, η ταυτότητα των μετόχων της Τράπεζας της Αγγλίας παραμένει μυστική. Ρώτησα εάν αυτό είναι αντίθετο προς την, τον κοινοτικό νόμο και αν το νέο σώμα θα μπορεί να αποκαλύψει τα ονόματα των, μετόχων ε, της Τράπεζας της Αγγλίας. Η Κομισιόν θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι νόμοι της να έχουν συνέπεια διαφάνεια για όλες τις χώρες. Ε, Ευχαριστώ κύριε Μπάτεν για τους μη εγγεγραμμένους. Ο κύριος Μάρτιν ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ. Ωραία που είστε εδώ κύριε Επίτροπε σήμερα. Οι προσπάθειες που έχετε κάνει τα χρόνια όπου ήσασταν αρμόδιος για τα θέματα αυτά έχουν αναγνωριστεί. Γνωρίζετε βέβαια και εσείς ο ίδιος ότι ο δρόμος ακόμα είναι μακρός. Δύο σχόλια. Νομίζω ότι είναι σωστό οι άνθρωποι που ε, γίνονται δεχτοί να κρίνονται εφόσον κάνουν δηλώσεις που δεν είναι ε, αληθείς και θα πρέπει να είναι δυνατόν να υφίσταται και κυρώσεις. Το δεύτερο είναι ποιος εκπροσωπείται. Γνωρίζετε και από, την, από τομέα της οικονομίας εκεί υπάρχει και ίδιο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανοιχτεί στους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών βλέποντας τα αποτελέσματα στον τομέα των οικονομικών σκανδάλων και της οικονομικής κρίσης βλέπουμε ότι οι συμβουλές που έχετε λάβει δεν ήταν ορθές και εδώ χρειάζεται δουλειά. Ευχαριστώ κύριε Μάρτιν. Για δύο λεπτά η κυρία Ζαμπόρσκα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φιλελεύθερους που άνοιξαν αυτό το θέμα, τη συζήτηση. Το πρόβλημα των εμπειρογνωμένων δεν περιορίζεται στην οικονομία. Σε άλλους τομείς η Κομισιόν δεν τήρησε τους κανόνες της αμεροληψίας, της διαφάνειας και οι ομάδες εμπειρογνωμόνων δεν εκπροσωπούν όλους τους πολίτες. Πρώτα απ' όλα ε, η οικογένεια περιλαμβάνει έναν άνδρα, ε, μια γυναίκα και παιδιά και ε, εκπροσωπεί μεγάλο τμήμα του πληθυσμού του ευρωπαϊκού αλλά έχουμε στην οικογενειακή πλατφόρμα τα λόμπι των γυναικών που προσπαθούν να υπονομεύσουν αυτό το μοντέλο της οικογένειας. Η Κομισιό απορρίπτει τις οργανώσεις της γυναικείας που αντιτίθενται σε ε, στην μονομερή θεωρία της οικογένειας. Έχουμε επίσης την υπηρεσία των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που χρηματοδοτείται από την Κομισιό οι εμπειρογνώμονες έχουν μια υποκειμενική ατζέντα χωρίς να έχουν μια αντικειμενική προσέγγιση. Ένα άλλο παράδειγμα ε, είναι αυτό το Κοινοβούλιο επίσης και ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει αποκλίνει από τις γνωμοδοτήσεις σχετικά με την θρησκευτική ελευθερία επειδή προετοιμάστηκε από λόμπι οργανώσεων που είναι υπέρ των αμβλώσεων. Νομίζω ότι ακόμα ε, και οι υπηρεσίε εμπειρογνωμόνων ε, ε, τα, όταν προτιμούν τα συμφέροντα ιδιωτών από το γενικό συμφέρον πρέπει να διαλύονται. Μπορώ να δώσω πάρα πολλά παραδείγματα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι συμμερίζομαι την ερώτηση που τέθηκε στην Κομισιό. Ζητώ από την Κομισιό να ανοίξει όλα τα παράθυρα στα γραφεία των εμπειρογνωμόνων, διότι εκεί ο αέρας, η ατμόσφαιρα δεν είναι καθαρή. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την οικονομία. Ευχαριστώ κυρία Ζαμπόρσκα για δύο λεπτά. Η κυρία Ματιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εργασία διαβούλευσης και συζήτησης με τους, με τους πρέπει να είναι άμεμπτη ως προς τη διαφάνεια διότι είναι μια επικίνδυνη δουλειά. Διότι ανάλογα με τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα του καθένα εμπειρογνώμονα πρέπει να γίνεται η επιλογή χωρίς να αντιβαίνει στα κοινά συμφέροντα. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη επίσης η αντιπροσωπευτικότητά τους αλλά και η δυνατότητα αντίθεσης. Πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν αντίθετα συμφέροντα μεταξύ τους. Θα έπρεπε λοιπόν στις διάφορες συναντήσεις να γίνεται συνάντηση μεταξύ όλων αυτών απέναντι στο ευρύ κοινό. Οι εργασίες των εμπειρογνωμόνων, των ομάδων εργασίας των εμπειρογνωμόνων δεν θα πρέπει να οδηγούν σε τελεσίδικα αποτελέσματα για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελεσματική εργασία θα πρέπει να προσωτεριστεί η Κομισιόν το Κοινοβούλιο ούτω ώστε να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της συνθήκης όλοι είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Ευχαριστώ κυρία Ματιέ για δύο λεπτά ο κύριος Γιακολίνο. Ευχαριστώ. Στην καθημερινή μας κοινοβουλευτική ζωή εμείς ε, διαπιστώνουμε ότι τη προστιθέμενη αξία των εργασιών μας ε, ε, προσδίδεται και από την πρόσθετη πληροφορία που διαθέτουμε. Και αυτό το πετυχαίνει η Επιτροπή με εξωτερικούς ανθρώπινους πόρους οι οποίοι δουλεύουν προς τον τομέα της πληροφόρησης βιομηχανικές, πολιτικές κλπ. Αλλά η πολιτική όμως παραμένει στα χέρια των πολιτικών. Αυτές είναι οι επιλογές, σίγουρα είναι επιλογές οι οποίες εμπίπτουν σε ομάδες εμπειρογνωμόνων με υψηλό επίπεδο κατάρτισης και επαγγελματισμού και πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική ισορροπημένα των όσων εκφράζουν. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να βρούμε διαφανείς διαδικασίες και αποτελεσματικά μέσα που θα επιτρέπουν στην Κομισιό να, κρατάει το ρόλο της υποστηρι... με την υποστήριξη αυτών των ομάδων εμπειρογνωμόνων που πρέπει να είναι αυτόνομοι ή ανεξάρτητοι. Ξέρουμε βέβαια ότι κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το σχέδιο του 2010 είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα πράγματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Η αξιοπιστία των εμπειρογνωμόνων εξαρτάται από την αυτονομία τους και από την ικανότητά τους να δέχονται τις πολιτικές αποφάσεις. Το Κοινοβούλιο αλλά και άλλες μέσα στο Κοινοβούλιο οι δυνατότητες ε, διαφάνειας μπορούν να πλωστευθούν όπως επίσης και στα πλαίσια της πρόσβασης του Ιντερνετ. Η διαφάνεια, η διαφάνεια όμως δεν θα πρέπει να γίνεται χωρίς να είναι αναγνωρίσιμος αυτός που έχει την πρόσβαση. Επίσης θα πρέπει να γίνει καταγραφή και των ομάδων πίεσης, των λόμπις. Όταν ο εμπειρογνώμονας είναι αξιόπιστος τότε είναι χρήσιμος. Η απόφαση όμως παραμένει στον πολιτικό που τον προσλαμβάνει. Ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο. Catch Ο κύριος Πάσκα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξέτασε το έγγραφό της για το έργο των εμιγρών ομόνων. Όλοι έχουμε επενδυμένα συμφέροντα για την βέλτιστη δυνατή λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης με τρόπο διαφανή. Με τον ίδιο διαφανή τρόπο πρέπει να ε, συντίθενται και τα συμβουλευτικά αυτά όργανα. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να ε, διορίζει τους εμπειρογνώμονες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόσφατα, ως παράδειγμα, είχαμε το παράδειγμα μάλλον του οργανισμού φαρμάκων όπου τα πράγματα δεν πήγαν όπως έπρεπε. Θα έπρεπε να κάνουμε μια συντονισμένη προσπάθεια ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι ομάδες εμπειρογνωμόνων και συμβούλων ώστε αυτές οι ομάδες ε, εμπειρογνωμόνων και συμβούλων είναι απολύτω αντικειμενικές και πρέπει να ληφθούν μέτρα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Πάσκα. Ο κύριος Όμπερ Μάιερ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Ο Επίτροπος κύριος Μπαρνιέ δέχτηκε ότι η σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι πάντοτε ισορροπημένες. Σε ορισμένες ομάδες εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνονται για παράδειγμα περισσότεροι εμπειρογνώμονες ε, του, της ομάδας ε, ε, του κλάδου των χρηματοπιστωτικών από ότι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι σοβαρά αυτά. Με τέτοιο τρόπο δεν διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια. Το ίδιο συμβαίνει και στον Οργανισμό ε, Ασφάλειας Τροφίμων που βασίζονται σε συμβουλές εμπειρογνωμόνων που όμως είναι προφανές ότι διαπλέκονται με ε, επιχειρήσεις που παράγουν τα προϊόντα αυτά. Χρειάζεται λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι μια νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία παράγεται βασισμένη σε αυτές τις συμβουλές είναι επικίνδυνη για τον πολίτη. Ευχαριστώ κύριε Βερμάιερ. Κύριε Πίτροπε έχετε άφθονο υλικό για να απαντήσετε. Ευχαριστώ αξιότιμα μέλη. Νομίζω ότι ε, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η συζήτηση και θα ήταν πάρα πολύ καλό να έχουμε ένα ε, μνημόνιο, θέλετε, ένα σημείωμα για το ιστορικό αυτό του θέματος. Βεβαίως η Επιτροπή σημείωσε όλες τις καλές ιδέες και συμβουλές που θα αυξήσουν τη διαφάνεια. Θυμάμαι τα το 2005 όταν αρχίσαμε μια πρωτοβουλία διαφάνειας που περιλάμβανε το θέμα των ομάδων εμπειρογνωμένων. Και ήταν κατά κάποιο τρόπο το παιδί μου αυτό, όπως θυμήθηκε ο κύριος Μάρτιν. Βεβαίως, ε, υπήρξε μεγάλη εξέλιξη σχετικά με το θέμα αυτό. Έχουμε ιστοσελίδες, έχουμε πληροφορίες, αλλά δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρείτε ότι οι εμπειρογνώμονες λαμβάνουν αποφάσεις. Δεν λαμβάνουν υποφέσεις, συγκρούονται μεταξύ τους, έχουν αντικρώμενες απόψεις σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, παραδείγματο χάρη. Υπάρχουν διαφορετικές ομάδες εμπειρογνωμένων, των οποίων η αποστολή διαρκεί μερικούς μήνες και έχουν ευθύνη είχαν επίσης και για την ασφάλεια όλα τα θέματα, όλες οι πληροφορίες ε, για τις ε, διάφορες επιδείξεις ε, ήρθαν στο γραφείο μου. Έγινε μία πρόσφατα για την κατάργηση των επιδοτήσεων στους παραγωγούς. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις επιτρόπων, οι απόψεις των επιτρόπων, των βουλευτών, τα κράτη-μέλη, οι κυβερνήσεις, οι εμπειρογνώμονες δεν λαμβάνουν αποφάσεις. Βεβαίως είμαι υπέρ μιας μεγαλύτερης διαφάνειας και είναι σαφές ότι <clears throat> μερικοί εμπειρογνώμενες είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Πάρα πολλές ομάδες συστάθηκαν αλλά διαλύθηκαν λίγο καιρό μετά διότι δεν μπορούσαν να δώσουν γνωμοδότηση, να γνωμοδοτήσουν διότι είχαν αντίθετη γνώμη μεταξύ τους. Έχουμε αυτό το μητρό διαφάνειας που θεωρώ ένα μεγάλο επίτευγμα, διότι οι εμπειρογνώμενες και οι σύμβουλοι υπάρχουν παντού. Κανένας πολιτικός δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς συμβούλους. Οι πολιτικές ομάδες είναι σύμβουλοι, έχουν διαφορετική προσέγγιση και ε, για μια πολιτική απόφαση ακολουθούμε μία θέση, τη μία ή την άλλη. Βεβαίως πολλές φορές οι εμπειρογνώμονες συμβουλεύουν για την υιοθέτηση μιας θέσης και απόφασης, αλλά δεν λαμβάνουν αποφάσεις. Έχουμε τους επιτρόπους, τους πολιτικούς, ε, τους ευρωβουλευτές, όπως σε κάθε δημοκρατικό σύστημα. Και βεβαίως ε, πάρα πολλά θέματα τέθηκαν για την σύνθεση τι πώς μπορεί να είναι εξισορροπημένη η σύνθεση, ποιος θα εκτιμήσει αν είναι εξισορροπημένη η σύνθεση των ομάδων. Κάθε συγκεκριμένη περίπτωση είναι διαφορετική ε, και από αυτήν ε, εξαρτάται η σύνθεση της ομάδας. Πολλοί θέλουν ε, να είναι μέλη των ομάδων εμπειρογνωμόνων για να λαμβάνουν αποφάσεις, αλλά δεν είναι αυτή η περίπτωση, δεν λαμβάνουν αποφάσεις οι ομάδες αυτές. Το 2005 θα θυμάστε ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό, αλλά παρέμεινε ασαφές από τότε. Η Κομισιόν επέφερε σημαντικές αλλαγές στην όλη εξέλιξη του θέματος μαζί με αυτόν το Κοινοβούλιο, ε, το σχετικά με το Μητρό ε, που έχουμε για τους εκπροσώπους και αυτό ε, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Έχουμε πολλά λόμπι, λόμπι εδώ, λόμπι στην Επιτροπή πόσο μεγάλη είναι η επιρροή τους ε, και το θέμα της σύνθεσης έχει σημασία. Ας συζητούμε το θέμα αυτό, αλλά να μην υποτιμούμε τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο. Και τώρα μπορείτε να πάτε για καφέ μέχρι τις 12 ακριβώς, οπότε θα αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ.